Ε, υπάρχει καμία αντίρρηση στην διάσκεψη των Προέδρων των ε, Επιτροπών στις τέσσερις συστάσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ να μην αντιταχθεί σε μια κατεξουδότηση πράξη. Εάν μέσα σε 24 ώρες καμία πολιτική ομάδα ή κανένας αριθμός βουλευτών ε, με βάση το κατώτατο όριο δεν θέσει αντιρρήσεις, τότε οι συστάσεις αυτές θα εγκριθούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα ψηφιστούν οι συστάσεις αυτές. Οι συστάσεις αυτές υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Και τώρα πάμε στη